Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τις ε, εργασίες μας της ε, Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, μπορούμε νομίζω να εγκρίνουμε την ημέρη αδιάταξη. Λάβατε γνώση των πρακτικών της συνεδρίασης της 1ης και της 2ης Απριλίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν μπορούμε να, τις εγκρίνουμε, να τα εγκρίνουμε. Υπάρχει και τα πρώτα πρακτικά της συνεδρίας των συντονιστών της 1ης Απριλίου. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση ούτε από αυτού μπορούμε να τα εγκρίνουμε και ερχόμαστε τώρα στην έκθεση που ε, μου αναθέσατε. Ήταν μια τιμή για μένα. Αυτό το σχέδιο κανονισμού δημιουργεί νομική βάση που επιτρέπει στο Μένο Βασίλειο να συνεισφέρει στον κοινοτικό προπολογισμό του 2019 και βεβαίω ε, οι δικαιούχοι που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στον Ευρωπαϊκό Βασίλειο, μπορούν να συμμετάσχουν ε, στα σχετικά προγράμματα. Το σχέδιο κανονισμού θα εφαρμοστεί μόνο εφόσον ε, αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς συμφωνία. Τώρα θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα φύγει. Εν πάση προς το Κοινοβούλιο θα πρέπει σήμερα να εκφράσει τη γνώμη του για το σχέδιο πριν εγκριθεί και από το Συμβούλιο ομοφόνος θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το κείμενο αυτό την ερχόμενη εβδομάδα μετά την ψηφοφορία εδώ σήμερα. Έχετε λάβει γνώση αυτής της έκθεσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πήρε μία ακόμα προθεσμία για μία υποθετική αποχώρηση, την παραμονή του Halloween, έτσι είναι η προθεσμία αυτή. στο τέλος την πραγματικότητα της ε, ε θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουμε νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Πάντως η οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση συχνά δίνει τον τόνο στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε, νομίζω, από την συνάντηση ονομαστική ψηφοφορία Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας για να δοκιμάσουμε πρώτα. Εγώ δεν έχω την κάρτα μου, αλλά θα σηκώνω το χέρι και προφανώς ε, είμαι υπέρ ε, της έκθεσης αυτής. Θέλω να δω αν μπορείτε να ψηφίσετε όλοι σε αυτήν την ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Ψήφισαν 15 υπέρ, γιατί είναι και δική μου ψήφο, μία ψήφος κατά και, και μία αποχή. Υπάρχουν άλλα θέματα για σήμερα το πρωί. Μάλλον όχι. Θα τα πούμε λοιπόν στο Στρασβούργο. Όχι, συγγνώμη. Η κυρία Γκρέσλε, συγγνώμη, ναι. Γνωρίζω ότι σας χρωστάω ένα μπουκάλι σαμπάνια, έτσι δεν το ξεχνάω. Ναι, ακούστε εκτός συνεδρίας αυτά. Εγώ πιστεύω ότι το μενό, Βασίλειο θα μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η οικονομική πραγματικότητα είναι ισχυρότερη από το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα χρειαστεί ίσως κάποτε το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα να υπάρξει ε, για να μπορέσει να γίνει μια μεγάλη δύναμη Ευρώπη. Ε, λοιπόν, θα τα πούμε στα σχόλια την επόμενη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε και εδώ βεβαίω στι 5 Ιουνίου. Όταν λέω εδώ, ενώ στι Βρυξέλλε, έτσι γενικά, όχι απαραίτητα Στην την αίθουσα, για μια έκτακτη συνεδρίαση που θα μα επιτρέψει να λάβουμε γνώση του σχέδιου προπολογισμού για το 2020 για όσους από εσάς είναι υποψήφοι και θα εκλεγούν βέβαια προφανώς. Ξεκινάει έτσι μια ενδιαφέρουσα περίοδος. Για όσους από εμά, ε, όπως εγώ, ε, θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμού, θα είναι μια συγκινητική στιγμή όπως και να το κάνουμε. Ελπίζω να είμαστε λοιπόν πολλοί εδώ στις 5 Ιουνίου. Ε, θα πιούμε και κάτι, ένα ποτήρι του αποχαιρετισμού και να ευχηθούμε τα καλύτερα στους υποψηφίους. θα μπορέσουμε πια να γιορτάσουμε την εκλογή τους βέβαια, πέρας ψηφοφορίας και πέρας της συνεδρίασης.